Good Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια ακρόαση για ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα μιλώντας για την ευρωπαϊκή πολιτική και τα τεστροτικά ταμεία, πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές ε, των ίσων ευκαιριών, της όρτας μεταξύ των δύο φύλων και αποφασίσαμε να υποβάλουμε μια έκθεση για να μπορέσουμε να συλλέξουμε βέλτιστες πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και προτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα πλαίσια της ανάπτυξης των πρωτοβουλίων αυτών. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην ε, συνάδελφο την κυρία Μούντι, η οποία είναι η συγγύτρια υπεύθυνη για την ε, γνωμοδότηση αυτή και στη συνέχεια θα μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες να θα ακούσουμε τις δικές τους απόψεις και βεβαίως αν υπάρχει χρόνος θα γίνει και μια συζήτηση. Για να μην χάνουμε χρόνο ακριβώς και να ξεκινήσει η ακρόαση θα δώσω το λόγο αυτής αμέσως στη συνάδελφο Κλέρ Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, σχετικά σύντομη για να μπορέσουμε να ακούσουμε κυρίως τους εμπειρογνώμονες που είναι εδώ σήμερα το απόγευμα, διότι το πιο σημαντικό είναι να γίνει μια συζήτηση ενημερωμένη, στοιχειοθετημένη στο Κοινοβούλιο και γενικότερα για τα ωφέλη των γυναικών από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση και η ακρόαση η σημερινή αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο γενικότερα, δεν αφορά δηλαδή μια συγκεκριμένη μορφή χρηματοδότησης. Κάνουμε πολλά καλά πράγματα για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει νομοθεσία για την απασχόληση, ε, νομοθεσία για την ισότητα, όμως χρόνο με το χρόνο υπάρχουν υπάρχει σημαντικό αντίκτυπο από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Πρέπει αυτό να τον μετρήσουμε τον αντίκτυπο. Να δούμε πού τα πράγματα πάνε καλά, πού δεν πάνε καλά, πού ο αντίκτυπο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, τόσο θετικό όσο θα θέλαμε και βεβαίω από εκεί πέρα τι μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα, κάποια στιγμή ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα είναι gender mainstream. Ε, αυτό είναι μια πραγματικά απτή δράση της Ένωσης, την οποία πρέπει να επιδιώξουμε ε, ακόμα πιο έντονα στο μέλλον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην Πρόεδρο για να ακούσουμε τους Σας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μούντι. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στο πρώτο πάνελ αξιολόγηση της ισότητας των δύο φύλων, πώς ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης ε, συνεισφέρει στη μείωση των ανισοτήτων. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Diane Μπάνιαν από την Bristol Women's Voice. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε για αυτή την παρουσίαση, πρέπει να πω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια προσπάθεια της εξέτασης του αντικτύπου για την πόλη μου, μετά και την, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν μια δουλειά που κάναμε με θετικό σκοπό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Το δίκτυό μας ε, αποτελείται από πολλές οργανώσεις γυναικών στο Μπρίστολ. Το Μπρίστολ είναι μια πόλη 400.000 περίπου ανθρώπων στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι ένα δίκτυο πολύ διαδεδομένο στην πόλη, πολύ διευρυμένο. Προσπαθούμε λοιπόν για να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία να έχουμε ένα όσο γίνεται πιο διευρυμένο δίκτυο. Το Μπρίστολ, το Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχείο του Bristol έχει δεχτεί πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ ε, από το 2005 στο 2015 ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τα δύο πανεπιστήμια έχουν λάβει 23, 23 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Horizon στην, στον Εμένο Βασίλειο και υπάρχουν επίσης 66 εκατομμύρια ε, από τα διαθροτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν στην πόλη μας στην περιοχή, καλύτερα, στην περιφέρεια. Να δώσω κάποια παραδείγματα με χρηματοδότησης που, από τα οποία αποφελήθηκαν συγκεκριμένα οι γυναίκες. Ε, πολλές φορές ε, δεν είναι από τα πανεπιστήμια στην πρώτη γραμμή, δεν ήταν η βασική εταίρη, αλλά ήταν εταίρη. Ε, και αυτή η συνεργασία ήταν εξαιρετικά επωφελής. Ήταν από τα πιο θετικά στοιχεία. Η συντονισμένη δράση κατά ε, της ε, βίας, της ενδοκογενειακής βίας ε, μας έδωσε υλικό ε, για τους, κατα, τους καταρτιζόμενους και για αυτούς που θα ασχοληθούν στο μέλλον με το να εντοπίζουν ποιες γυναίκες έχουν πέσει θύματα ενδοκογενειακής βίας. Ε, έχουμε εκατοντάδες, έχουν καταρτήσει εκατοντάδες Συμβούλου ε, για το ζήτημα αυτό. Είχε πραγματικά απτά αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι η κοινοτική μας οργάνωση στο Μπρίστολ αλλά και στον Εμένο Βασίλειο γενικότερα ασχολείται με κοινότητες που έχουν υποστεί ε, υπήρξε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Εργαστήκαμε με νέους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, τους οποίους ε, προσπαθήσαμε να ε, καταστήσουμε πολέμιους, αν θέλετε, αυτής της πρακτικής στις κοινότητές τους. Είχε μια ευρεία εμβέλεια αυτό το πρόγραμμα. Μία νεαρή γυναίκα που συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα μάλιστα κάποια στιγμή μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη για την εμπειρία της, ε, ε της ε, καταπολέμησης, ε, της μάχης κατά της κλειτοριδεκτομής. Είχαμε ένα άλλο καινοτόμο πρόγραμμα με επαγγελματίες του τομέα της ποινική δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά άτομα τα οποία έχουν ζήσει περιπτώσεις ενδοκονομικής, βία βίας και που προσέφηγαν στη δικαιοσύνη. Ήταν λοιπόν ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση των επαγγελματιών για να καταλάβουν την περιπλοκότητα και τη δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα όταν έχει, να, έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα πάλι που βασίζεται στις τοπικές κοινότητες, πάλι που αφορά νέους ανθρώπους είναι μια εφαρμογή για να υπάρξει υποστήριξη από, την ευκαιρία, από τις εμπειρίες των νέων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και την πίεση που δημιουργούνται μέσα στις σχέσεις που δημιουργείται μέσα στις σχέσεις είναι ένα πρόγραμμα που αφορά κυρίως νέους ανθρώπους και τέλος οι επιπτώσεις των εργασιών με άντρες οι οποίοι ε, είναι βίαιοι στην ιδιωτική του ζωή με τον ε, σύντροφό τους ε, και από εδώ προέκυψαν κάποια παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για το τι λειτουργήσε και τι όχι. Είχαμε δηλαδή κάποια αποτελέσματα στοιχειοθετημένα, κάτι που πάντα είναι χρήσιμο. Σε σχέση τώρα με άλλα προγράμματα, το Progress για την κάλυψη του κενού, του χάσματος. Πρώτα απ' όλα εδώ εξετάσαμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων για τη μείωση των, της απόκλησης της αμοιβέ. Είχαμε κατευθύνσει γραμμέ για να υποστηριχθούν τα συνδικάτα αλλά και οι εργοδότε, οι εταιρείε για μια σειρά αποζητήματα τα οποία επηρεάζουν το θέμα ακριβώ της αντιμετώπιση ε, του χάσματος που υπάρχει μεταξύ, στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πώς δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό συγκεκριμένα. Εδώ το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αγγλίας ήταν ε, εταίρος στο όλο εγχείρημα. Αυτά έχουν πλέον ενσωματωθεί μέσω της, ε, ε των οργανώσεών μας στις πρακτικές ε, στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης ε, μια πρωτοβουλία της, της Γενικής της Δικαιοσύνης για τις ε, ε με, γυναίκες μετόχους που ζητούν ισότητα των δύο φύλων. Θέλουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε εδώ τη διαδικασία των μετόχων για να, που θα μπορούσαν να πιέσουν τις εταιρείες για να δώσουν πληροφορίες για το ποιες δράσεις αναλαμβάνουν για να αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και γενικότερα σε υψηλόβαθμες θέσεις και η βέλτιστη πρακτική που προέκυψε από εκεί έχει χρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο για να μπορέσουμε ακριβώς να πιέσουμε κάποιες εταιρείε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα, τα, τα διαδοτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων, ε, αυτό δεν αφορούσε άμεσα απευθείας τις γυναίκες, υπήρχε όμως η απέτηση να ασχοληθούν με το ζήτημα της άντρας των δύο φύλων, ε, είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η χρηματοδότηση που έχουν, έχει να κάνει με τις δεξιότητες, με την απασχόληση. Εδώ έχουμε απλά κάποια παραδείγματα. Ένα από αυτά ήταν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, να οργανωθούν μαθήματα γλωσσών για ανθρώπους που τα αγγλικά δεν είναι η μητρική τους και δυσκολευόντουσαν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία Αυτά τα μαθήματα γλωσσών θα μπορούσε ταυτόχρονα να να συναδεύονται με φροντίδα των παιδιών. Ε, έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκες να παρακολουθούν το μάθημα ενώ υπάρχει φύλαξη των παιδιών τους. Ε, επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μπορούσε αυτό να ενσωματωθεί σε ένα σχολείο. Εν πάση περιπτώσει εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες το πρόγραμμα αυτό. Ε, το οργάνωσε το Ashley Housing Association ε, που οργανώνει και ε, ε, όπου συμμετέχουν μάλλον πολλοί αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα έχει γίνει δεκτό το πρόγραμμα για τη μετατροπή των υπάρχων δεξιοτήτων ε, αυτό το πρόγραμμα προχωράει μέσω των σχολείων και αναπτύσσεται από εθελοντικές οργανώσεις ε, στις τοπικές κοινότητες αυτό οργανώθηκε από τις ε, γυναίκες πρόσφυγες του Μπρίστολ και συνεισέφερε έτσι ώστε οι δεξιότητες που υπάρχουν στους ανθρώπους αυτούς να αναγνωριστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατροί, μηχανικοί, οδοντίατροι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους, τα προσόντα τους και να μπορέσουν ε, να περάσουν από μια χαμηλά αμοιβόμενη εργασία, άνθρωποι δηλαδή που είχαν δεξιότητες και δουλεύαν ως ε, ε οικιακό προσωπικό μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά τις δυνατότητε τους. Από εκεί και πέρα είχαμε και το πρόγραμμα ε, για τις ε, γυναίκες που εργάζονται στο τεχνικό σκέλος ε, των κινηματογραφικών ταινιών καθώς ε, και στον τομέα της οικοδομής. Είναι προγράμματα τα οποία προχωρούν με διάφορους τρόπους τα διδάγματα που προκύπτουν από τα προγράμματα αυτά περνούν και στην επόμενη γενιά των σχετικών προγραμμάτων. Πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικό η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων να αποτελεί οριζό, να έχει ένα οριζόντιο χαρακτήρα, να υπάρξει mainstreaming δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τον, το Horizon, αυτοί που εργάζονται στο πρόγραμμα Horizon, η απέτηση να υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στις ε, ε, ομάδες έρευνας, ε, να, υπάρχουν, να υπάρχει τουλάχιστον 40% εκπροσώπηση και 50% στις ε, συμβουλευτικές ομάδες, πραγματικά θα αλλάξει τα πράγματα στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να υποτιμήσουμε ως μέσο για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στο επιστημονικό πεδίο, στο τεχνολογικό πεδίο, το μαθηματικά, όπου οι γυναίκες εκπροσωπούνται. Αυτό το mainstream για τις ευκαιρίες πρέπει να προβλέπεται και ε, στο, ε, στα ταμεία, τα διαθροτικά. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης να το λάβουν υπόψη τους αυτόν, να καταλάβουν ότι δεν πρέπει οι γυναίκε να θεωρηθούν απλά ω δικαιούχοι ε, κάποιων ε, δικαιωμάτων ή υπηρεσιών, αλλά πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίση, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι σημαντικό για μα τον Πρίστολ. Είμαστε μεταξύ των ε, αυτών που έχουν υπογράψει τη χάρτα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην τοπική ζωή είναι κάτι το οποίο ε, παρακολουθείται από το EIG. Έχουμε πάνω από 1.200 ε, υπογράφοντες ε, συμβαλόμενους σε αυτή τη σύμβαση. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο βάλει των πρακτικών, γίνονται εκδηλώσεις όπου μπορούν μπορεί ο καθένα να στείλει τι καλέ πρακτικέ για διάφορε πτυχέ τη χάρτα. Προσπαθούμε να έχουμε εκπροσώπηση 50-50 στα τοπικά συμβούλια και το φτάσαμε στο 43%, όχι στο 50%, στο 43%, σημαντική άνοδος όμως. Ε, από εκεί και πέρα τα δεδομένα τα οποία ε, προκύπτουν από το Ινστιτούτο είναι εξαιρετικά χρήσιμα διότι είναι αυτά ακριβώς τα στοιχειοθετημένα, αξιόπιστα δεδομένα για να μπορούμε να πούμε ότι ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε ε, εργαλεία, βέλτιστη πρακτική, βέλτιστες πρακτικές, ε, ευαισθητοποίηση του κοινού. Ήθελα επίσης να μιλήσω για το πλαίσιο προγραμματικής συνεργασίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, έχουμε, έχουμε εργαζόμαστε στα πλαίσια μιας, ενός, ένα προγράμματος, ενός προγράμματος κοινούς χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης στα πλαίσια και ε, της ε, εταιρικής σχέσης, της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Θέλουμε και εδώ βεβαίως να έχουμε στοιχεία ε, αξιόπιστα εξετάζοντας τα ζητήματα που ε, εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετέχουν σε εκλογικέ διαδικασίες και στο τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, ε, να εξετάσουμε και εδώ τι βέλτιστες πρακτικέ Είναι ένα θέμα. Έγινε έρευνα λοιπόν ε, σε μια σειρά από χώρε σε οικονομικό, σε κοινωνικό επίπεδο. Ε, είχαμε συνεντεύξεις με γυναίκες εκλεγμένες, αυτές που τα κατάφεραν, αυτές που δεν τα κατάφεραν η σχετική έκθεση θα δημοσιευτεί, θα παρουσιαστεί μάλλον ε, το Δεκέμβριο. Τα στερεότυπα, η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι τα δύο βασικά ζητήματα. Υπάρχει ένας κατάλογος συστάσεων που έχει προκύψει και για την κάθε χώρα ξεχωριστά και για την περιοχή αυτή γενικότερα. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένες συζητήσεις για το τι θα μπορούσε να ελοποιηθεί από όλα αυτά. Είναι ένα σημαντικό μέρος πάντως και αυτό των εργασιών μας. Και τέλος, σε ό,τι αφορά, θα ήθελα να πω ότι με τα εργαλεία και με τη θέλησή μας μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Βεβαίως η πολιτική βούληση είναι το πιο σημαντικό, αλλά υπάρχει μία απέτηση να συμβεί αυτό. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για ένα τομέα, ένα κλάδο ε, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει σοβαρά, παίρνει στα σοβαρά, τόσο σοβαρά ώστε να την χρηματοδοτεί επαρκώς. Είναι όμως σημαντικό να υπάρχει και παρακολούθηση, αποτελεσματική παρακολούθηση, διότι ο τελευταίος γύρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ηνωμένο Βασίλειο υποεκπροσωπήθηκε σε ό,τι αφορά τις, τις γυναίκες δικαιούχους. Και ο επόμενος γύρος ε, θα έχει τις ίδιες απαιτήσεις. Όχι μόνο, μόνο λοιπόν παρακολούθηση, αλλά και να λαμβάνουμε αποτελεσματική δράση. Αυτά είναι δύο ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Μπάνιεν. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα, τα οποία αναδείξατε και με βέβαιο ότι στη συνέχεια όσα είπατε θα προκαλέσουν ερωτήσεις αλλά και συζήτηση. Και όσον αφορά αυτό το οποίο μας είπατε στο τέλος, έχω και εγώ μια ερώτηση την οποία θα σας υποβάλω. Όμως, τώρα να πάμε ε, στην ε, επόμενη ομιλητριά μας, την κυρία Ντισάρτσινα, η οποία είναι εμπειρογνώμων του ε, Ιδρύματος για την Ισότητα των Φίλων στην ε, Ιταλία. Θα την ακούσουμε και κατόπιν να προχωρήσουμε. Κυρία Σάρτσι, να έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ και την κυρία Μούντι, την συγκίτρια και την κυρία Φαρέντσα για την ε, πρόσκλησή της. Για μένα είναι τιμή να παρίσταμε εδώ στη συνάντηση Επιτροπής των Γυναικείων Θεμάτων στο Κοινοβούλιο γιατί έχει ιστορική σημασία. Είναι θέμα οικοδόμησης της Ευρώπης αυτή η πολιτική των ίσων ευκαιριών και όλα αυτά τα έχουμε αναλύσει τι είναι μεταξύ 79 και 84 που δημιουργήθηκε και άρχισε την πορεία της αυτή η Επιτροπή σε σχέση με όσα γίνανε για την ε, επεξεργασία μιας στρατικής ίσων ευκαιριών. Έχουμε ε, αρχεία, παλαιά έγγραφα, συζητήσεις, ολομέλεια και όλα αυτά έδειξαν για το πώς εκείνη την πρώτη θητεία, η πρώτη επιτροπή ε, γυναικών έβαλε το λιθαράκι της Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Κάτι που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ε, σε όλες τις στρατηγικές. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 80. Και όπως είπε και η προλαλή σας, είπαμε ότι έχουμε το gender mainstreaming, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που ακολούθησε το δεκαετία του 90 με την συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα αυτό που συζητούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι έτσι θα ρίξουν άπλα το φως στο πώς συγκεκριμένα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει και να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με ε, τις ίσες ευκαιρίες. Πώς συγκεκριμένα μπορεί να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ζωή ανδρών και γυναικών παρά το ότι βρίσκεται σε βέβαια μια δύσκολη καμπή. Πρόκειται για ένα προβληματισμό επομένω που είναι πολύ επίκαιρο. Να δούμε όμως τι θα γίνει και για κάποια κενά που υπάρχουν, τις ε, επικρίσεις όσον αφορά τη δυνατότητα βελτιώσεις αυτού του προτσέσου. Πρόκειται επομένω για μια υπόσχεση, ένα καθήκον της Επιτροπής σας, μια δέσμευση. Και επίσης θα πρέπει να δοθεί νεόθεση στον διάλογο Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που γενικότερα ε, δεκαετία του 70 και 80 πέδωσε Κάρολ Επομένω, Επομένως, ε, ας αντιλήσουμε συμπεράσματα από αυτή την πρώτη ε, θητεία και την πρόεδρο τη Σιμών που και αυτή έδωσε αγώνες για τον ε, φεμινισμό στην Ευρώπη και τις ίσες ευκαιρίες. Οπότε έχουμε τώρα αυτό το ζεύγος που αφορά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τις ίσες ευκαιρίες. Θα πρέπει αυτό να το πλαισιώσουμε το δίδυμο και να το προωθήσουμε και να, επίσης να φροντίσουμε το πώς το δημοσιοπλαισιο πλαισιο πλαίσιο 2014-2020 να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων για την ισότητα ευκαιριών και ακριβώς όπως είπαμε τώρα θα πρέπει όλα αυτά να αναδείχνουν και με τα έγγραφα μέχρι το 2016-2019 υπάρχει σχετική στρατηγική. Έχει επομένω τους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετοχή στην ε, απασχόληση να μειωθεί η μισθολογική ανισότητα και να μην υπάρχουν τέτοιες ανισότητες αναφύλλω και οριζόντια και τομέα να καταπολεμηθεί η βία των γυναικών και να υπάρξει σεβασμός για τη γυναίκα παντού, σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια στρατηγική επομένως. Άρα αυτό το gender mainstreaming, η ενσωμάτωση του φίλου στις πολιτικές είναι πολύ σημαντική. Και βέβαια όσον αφορά την έγκριση του προπολογισμού, όπως είπε και η κυρία Μούντι, οδηγεί στο πρόγραμμα εργασίας για το 17. Οπότε και η υπόθεση της όντας των φύλων ελήφθη υπόψη στην κατάρτιση του προπολογισμού για την επόμενη χρήση του 17 και οι το και δύο ευρωβουλευτές Ιταλοί. Συχνά λέμε ότι χρειάζεται γνώση, γνώση συγκεκριμένη του τι σημαίνει η ενσωμάτωση διάσταση του φύλου. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τις ευκαιρίες χωρίς να τα λέμε με τα λόγου γνώσεως για αυτά τα θέματα. Άρα, έτσι θα πρέπει να γίνει η ένταξη γυναικών και ανδρών στην ε, αγορά εργασίας και η Virginia Γουλφ ε, είχε μιλήσει σχετικά με αυτό. Είχε γράψει τα ενδυστορήματά της και είχε πει ότι χρειάζονται λεφτά για μια γυναίκα. Χρειάζεται και να έχει το δικό της χώρο, το δικό της δωμάτιο για να συγγράψει. Να, πώς ήταν η κατάσταση και βλέπουμε ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία συμβάλλουν στο να υπάρχει περισσότερη πλαισίωση, ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ταμεία. Περίοδο 2014-2020 έχουμε τα διευθυντικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το πρόγραμμα που αφορά την απασχόληση και την ε, κοινωνική καινοτομία. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε ε, πώς λειτουργούν, πώς αποδίδουν αυτά τα ταμεία και να δούμε τι γίνεται με την χρηματοδότηση της εκταμιεύσης όσον αφορά την βοήθεια προς τις γυναίκες στην αγορά εργασία. Έχουμε τώρα το, το επενδυτικό ταμείο, τα ιδιωτικά ταμεία και ήταν πρώτο το κοινωνικό ταμείο που έκανε τις πρώτες εκταμιεύσεις προς χάρη των γυναικών στη δεκαετία του 70. Και τότε βοηθήθηκαν οι γυναίκες να έχουν επαγγελματική κατάρτιση, να μπουν στην αγορά εργασίας και έχουμε πάνω στα αλληλεπτικά προγράμματα με συνεργασία των κρατών μελών, ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περίοδο 2020 πρόκειται να έχουμε 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα βοηθήσουν την ισότητα των φύλων. Τώρα έχουμε το Ευρωκοινωνικό Ταμείο, τα Κοινωνικά Ταμεία, το Ταμείο Επενδύσεων. Αχ, σα τα λέω πολύ γρήγορα, συμπαθάτε με, λέει η ομιλήτρια. Οπότε είπαμε ότι το, Ευρωκοινωνικό Κοινωνικό Ταμείο, το Διορθωτικό Ταμείο, είναι τα ταμεία τα οποία μέχρι τέλος δεκαετίας του 1990 προωθούσαν, πλαισίωναν το mainstreaming. Και είχαμε επίσης και την πολιτική συνοχή της Ένωσης. Να θυμηθούμε ότι το mainstreaming αλλά και συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες εκταμιεύσεις γινόντουσαν και ακριβώ είχαν προβλεφθεί στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου. Επίσης έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία όλα αυτά συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι είχαμε πλαισίωση για την ανατροφή των ανηλίκων και επίσης αυτόν τον συγκερασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης είχαμε την ευρωπαϊκή κοινότητα της πρακτικής όσον αφορά το mainstreaming που ανέφερε στη το 2010 και 2014 και εκεί αναπτύχθηκαν διάφορε δραστηριότητε, ούτω ώστε η ενσωμάτωση τη υπόθεση τη πόθεσης της ε, ισότητας ε, προωθήθηκε μέσα από τα ευρωπαϊκά ταμεία σε σχέση με τους στόχους για το 2020. Και 70% ε, αφορά τις την κάλυψη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για σκοπούς απασχόλησης. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν κάποια πρότυπα όσον αφορά την ενσωμάτωση της ισότητας για όλα τα προγράμματα που προωθούνται από το Κοινωνικό Ταμείο. Και είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες για την υλοποίηση της ενσωμάτωσης της ισότητας αλλά το Γενικό Ταμείο πρόκειται πάρα πολύ αυτή την ε, υπόθεση. Το πώ θα γίνει η υλοποίηση αυτή τη αρχή. Τώρα, έχουμε και άλλα δύο ταμεία, τα οποία επίση συμβάλλουν ε, στην πλαισίωση της γυναίκας στην ε, αγορά εργασίας, το, το, Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και το Κοινωνικό Ταμείο επίσης. Όπως έλεγα στην αρχή τη ομιλίας μου, τα ευρωπαϊκά ταμεία βοηθούν για την ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασία, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη χειραφέτηση τη γυναίκα. Και σήμερα η προβληματική για αυτή τη χειραφέτηση ε, εστιάζεται στο ποιο είναι ο ρόλο των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Είναι χαμηλή η συμμετοχή 30 και 40% είναι η συμμετοχή σε αυτές τις θέσεις τις ε, διοικητικές. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει περισσότερη ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείε. Ε, στην Ιταλία έχουν γίνει βήματα πρόοδου με το νόμο 120 του 11 Ακριβώ αυτό έχει βοηθήσει για περισσότερη παρουσία σε ηγετικέ εταιρικέ θέσει των γυναικών. Και είπαμε ότι αυτό το, το δίδυμο, το δίπολο, τα μία ευρωπαϊκά και δικαιώματα της γυναίκας έχει ακόμα πολλή πορεία να κάνει για να οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Και υπάρχει τώρα ένα σημαντικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην παρουσία των γυναικών στα πανεπιστήμια. Πρόκειται για την εικόνα του, του αγωγού που έχει διαρροή. Βλέπετε εδώ πέρα σε αυτή την γραφική παράσταση τι γίνεται. Στην αρχή είναι περισσότερες οι γυναίκες αρχικής διαδρομής. Μετά όμως πέφτει η καμπύλη που αφορά τις γυναίκες και ανεβαίνει η καμπύλη που αφορά τους άντρες. Βέβαια έχουμε πολύ λιγότερες γυναίκες επίσης όσον αφορά τις θετικές επιστήμες. Και υπήρξε και μια σχετική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε επίση ένα πρόγραμμα πλαίσιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έρευνα και καινοτομία. Πρόκειται για μια πολιτική που έχει ελκύσει πολλούς κοινοτικούς πόρους. Ακριβώς το θέμα της συμμετοχής των γυναικών και στις θετικές ε, επιστήμες. είπαμε ότι ευτυχώς ε, συνεχίζεται αυτή η τάση και στο πρόγραμμα Ορίζον του 2020, σχετική πολιτική, και ε, είπαμε ότι θα πρέπει και σε έρευνα και καινοτομία να ισχύσει η ίδια τάση. Έχουμε συγκεκριμένα κονδύλια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων σε έρευνα και καινοτομία. Ε, αυτό ονομάζεται Jerry από τα αρχικά στα αγγλικά. Και έχουμε επομένω έτσι μια καινοτόμα προσέγγιση υπάρχει ένα βραβείο για κάποιο είδους ε, καινοτόμες ιδέες, ε, καινοτόμα ε, δημιουργήματα των γυναικών. Και υπάρχουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να δημιουργηθεί περισσότερη ισότητα σε παιδεία, σε εκπαίδευση, σε κατάρτιση και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, γιατί και εκεί υπάρχουν ανισότητες. Θα πρέπει επομένως να μειωθούν αυτές οι ανισότητες όσον αφορά τις βασικές καταρτήσεις, όσον αφορά την, την απουσία, την εγκατάλειψη του σχολείου. Επίσης να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και στην ανώτερη εκπαίδευση αλλά και στις θετικές επιστήμες. Επίσης να συμμετάσχουν περισσότερο γυναίκες στην επαγγελματική κατάρτιση γιατί οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες σε κάποιο είδου ε, μη αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα. Και υπάρχει πρόβλημα με την χρηματοδότηση, γιατί ακριβώς εκεί γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Επομένως, συμβάλλουν τα ευρωπαϊκά ταμεία στην υπόθεση της ε, ισότητας. Υπάρχουν και εδώ και βέβαια και κάποια στερεότυπα που θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Επίσης υπάρχει το έρασμος για όλους. Αλλά δεν λαμβάνεται εδώ υπόψη η υπόθεση της ισότητας των φύλων. Δεν υπάρχει κατάλληλη χρηματοδοτική πλαισίωση. Και έχω συνεργαστεί με το πρόγραμμα Ζαν Μονέ, το οποίο είναι τμήμα του έρασμος και γενικότερα το θέμα των ευρωπαϊκών ε, σπουδών, ε, γνώση δηλαδή των ευρωπαϊκών υποθέσεων και στο σχολείο αλλά και στο πανεπιστήμιο. Ε, και εκεί θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο η υπόθεση της ισότητας των ευκαιριών σε σχολείο και σε πανεπιστήμιο. Και έτσι θα επιτευχθούν πιο εύκολα οι στόχοι μας. Οπότε θα πρέπει οριζόντια να εξασφαλιστεί το gender mainstream. Γνώση της υπόθεσης ισότητα ευκαιριών μέσα από το έρασμος. Έτσι οι πολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες θα γίνουν πιο γνωστές. Να, πώς θα καταβληθούν και οι δυσμενείς διακρίσεις. Και μιλώ ότι υπάρχει έλλειμμα σε αυτό ακόμα και στον ανώτερο επίπεδο της ε, παιδείας. Τώρα υπάρχει και το θέμα της ε, βίας κατά των γυναικών και υπάρχει ένα σχετικό πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στην καταπολέμηση αυτής της ε, βίας. Ονομάζεται δικαιώματα, ισότητα και ιδιότητα του πολίτη. Για κάθε μορφή βίας υπάρχει ε, μια χρηματοδότηση από 440 εκατομμύρια ευρώ και 35% περίπου αφορά τα θέματα ισότητας και βίας κατά των γυναικών. Μια σειρά δράσεων θα μπορούσαν να γίνουν. Δραστηριότητα ανάλυσης, εκπαίδευσης και επίσης ε, εδώ συμβαίνουν πάρα πολύ και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όσον αφορά τώρα την πρόθεση των δικαιωμάτων γυναικών, εδώ υπάρχει κάποιο σχετικό ε, μέσο ή εργαλείο. Πώς τώρα θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτό το δίπολο Ευρωπαϊκά Ταμεία και ισότητα ευκαιριών. Τρία τινά είναι το ζουμί εδώ. Πρώτα-πρώτα περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη χρηματοδότηση όσον αφορά την ε, παιδεία, σχολείο και πανεπιστήμιο. Με το έρασμος επίσης. Ε, να καταπονήσουμε έτσι τις προκαταλήψεις και επίσης σε κάθε πρόγραμμα να υπάρχει χρηματοδότηση όσον αφορά το mainstreaming. Και αυτό να προβλέπεται από το δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Ακόμα και στο έρασμος είπαμε ότι δεν γίνεται αυτό. Να, ότι αυτή η διάσταση της όντας να ληφθεί υπόψη. Νομίζω όμως υποσέχθηκε το θέμα για τη χρήση του 2017 στον προπολογισμό. Τώρα έχουμε και κάποια καινούρια γενιά από project managers αυτοί προσέχουν τα θέματα ισότητας και μπορούν να λαμβάνουν την υπόθεση αυτή σε έργα και προγράμματα. Ο όλοι όσοι ασχολούνται με ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα γνωρίζουν τα της χρηματοδότησης, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την διάσταση, τη διάσταση του φύλου, το mainstreaming, gender mainstreaming. Οπότε, γι' αυτό σας λέω ότι έχω αυτές τις τρεις σκέψεις που θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε. Ό,τι τυχόν ρωτή θέλετε, ευχαρίστως να τις σχολιάσω. Ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε τον γύρο των ε, παρεμβάσεων. Κυρία Λεπιδίπη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ που έχει ασχοληθεί με αυτό το σημείο είναι η κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί. Οπότε μου είπε μήπως μπορέσω να σας πω συγχωρήσετε να την αντικαταστήσω και να λάβω τον λόγο αντί για εκείνη. Άρα, εκπροσωπώ τώρα την κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα στην Επιτροπή για τα θέματα των γυναικών έχουμε ασχοληθεί με ενεργό και παραγωγικό τρόπο χρόνια ούτω ώστε να γίνει μια αξιολόγηση του προϋπολογισμού για τα θέματα των φίλων Και έτσι τώρα ελήφθη υπόψη η διάσταση του φύλου. Ουσιαστικά σε κάθε βήμα της ε, έγκρισης και κατάρτισης αυτού και έτσι να υπάρχει κάποια προώθηση της υπόθεσης ισότητα των δύο φύλων. Επίσης, μέχρι τώρα αλλά και στο μέλλον, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακριβώς ε, υποσχέθηκε η κυρία Γιούροβα, έχουμε ασχοληθεί λέγω με την χρηματοδότηση των προγραμμάτων στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων του προϋπολογισμού εκδιάζονται κατά μία ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το κοινωνικό ταμείο και οι βασικές προτεραιότητες για το ΕΛΚ είναι το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο για να σημειωθεί ουσιαστικό βήμα προόδου για την ισότητα των δύο φύλων. Πρώτα-πρώτα ε, για την αγορά εργασίας, για το πώς θα υπάρξει εγγύηση του ότι θα υπάρχει μισθολογική ισότητα για ίση εργασία, ε, επίσης ε, εξασφάλιση της, του συγκερασμού του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο και αποκλεισμό των δυσμενών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Αυτά και άλλα, επομένως, έχουν απασχολήσει το ΕΛΚ. Και για λογαριασμό της κυρίας Ματέρεχο να σας θέσω δύο ερωτήματα. Βέβαια, ίσως τα έχετε καλύψει, ε, η κυρία Σαρτσίνα. Εσείς πού νομίζετε ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μπορεί να γίνει για να εξασφαλίσουμε οικονομική ανεξαρτησία σε άντρε και γυναίκες, δηλαδή μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο, το Κοινωνικό, τα Διαφορετικά κλπ. Μα είπατε για το Erasmus Plus. Τώρα τα υπεραπλουστεύω για να σας δώσω την εικόνα αυτών που θέλουμε και να δούμε το πώ το Erasmus Plus θα προσανατολιστεί περισσότερο προς το θέμα τη ισότητα. Άρα πώς μέσα από τον προπολογισμό μπορούμε να κάνουμε κάτι για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο, στην οικονομική ανεξαρτησία, να παρακάμψουμε δηλαδή, τα στερεότυπα και να καταπολεμήσουμε το τη μισθολογική ανισότητα. Επίσης, τι άλλο θα μπορούσατε να προτείνετε ότι μπορεί να γίνει για να πετύχουμε τους ε, στόχους μας, δηλαδή την άρση της ανισότητας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόντροβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντική και ο λόγος είναι ότι τώρα αντιμετωπίζουμε, έχουμε μπροστά μας διάφορες εκθέσεις που συνδέονται μεταξύ τους και γι' αυτό χρειαζόμαστε να ακούσουμε εμπειρογνώμονες. Ε, ευχαριστώ από καρδία τις ομιλήτης γιατί μας δίνουν παραδείγματα έρευνας όπου υπάρχει νόημα που μας παρέχουν τις ε, πληροφορίες που χρειαζόμαστε, όπως το Bristol Women's Voice. Πολύ αξιόλογη συμβόλη, όπως και η εμπειρία από την Ιταλία. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε εδώ τον Τσέχο ε, πραγματογνώμονα που θα μας ε, μιλήσει στη συνέχεια. Αν θέλουμε να αξιολογήσουμε αυτά τα προγράμματα, πώς λειτουργούν, πώς τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν να υποστηρίξουν την ισότητα των φίλων στα κράτη-μέλη, Στι διαφορετικέ περιοχές, τότε χρειαζόμαστε συγκεκριμένε πληροφορίες, ώστε να δούμε ποιε είναι οι τάσει. Μου άρεσε πολύ το παράδειγμα, ε, το παράδειγμα του ορίζοντα 2020, όπου χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο για να κινητοποιήσουμε και να εμπλέξουμε τις γυναίκες ε, στην έρευνα. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα για να διαδώσουμε. Η Ιταλίδα Μιλητρία αναφέρθηκε στην τύχη της οδηγίας που θα έπρεπε να μετριάσει να εξασφαλίσει ισότητα στη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Η τσεχική δημοκρατία έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Η Επίτροπος Γιώροβα το έχει κάνει κάτι πιο προσβάσιμο και, ε, παραδείγματος χάρη, η Τσεχία θα το εφαρμόσει δεν θα επωφεληθούν μόνο οι γυναίκες. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι είναι προς το συμφέρον ολόκληρη τη κοινωνία ώστε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό όλων των γυναικών, γιατί αλλιώ βγαίνουμε χαμένοι. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό και ελπίζω ότι οι γυναίκες ε, θα κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί περισσότερο. Το πρωί συζητήσαμε για την ε, έκθεση Πόρτασον, ήταν μια αξιολόγηση ε, της ισότητας στην περίοδο 2014-2015. Δυστυχώς αναφέρθηκε ότι η ισότητα των φύλων μειώνεται όσον αφορά τις προτεραιότητες και ότι μετατοπίζεται, ε, παραμερίζεται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνήσουμε, να αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν θέλουμε το θέμα αυτό της ισότητας των φίλων να γίνει δευτερεύον και να βγει από το επίκεντρο της προσοχής. Θέλουμε όμως παράλληλα να γνωρίζουμε και για ποιο λόγο οι πολιτικές αυτές δεν υποστηρίζονται όπως θα έπρεπε. Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσουμε, να εστιάσουμε περισσότερο σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ώστε να το κάνουμε πιο ελκυστικό ως θέμα. Η, κυρία Λεγκρίπ πρότεινε, μια, ε, την έκθεση για το συνταξιδοτικό χάσμα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το χάσμα. Τη χρειαζόμαστε αυτή την έκθεση και θέλω να σε ευχαριστήσω για την ε, έρευνα που διεξάγεται, για τα παραδείγματα που μας αναφέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε τις γνώσεις μας, ώστε να συνεισφέρει αυτή η Επιτροπή ε, στη δημιουργία νέων προτάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μόδη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τις ομιλήτριες μέχρι στιγμής για την πολύ σημαντική συνεισφορά τους. Η αναφορά που έγινε στα συγκεκριμένα παραδείγματα, αυτό όντως βοηθάει πολύ στο να ζωντανέψουμε και να δώσουμε έμφαση σε κάτι που δεν είναι απλά θεωρία, είναι πράξη. Το παράδειγμα του ορίζοντα 2020 όχι μόνο επειδή υπάρχει χάσμα στις δεξιότητες, αλλά υπάρχει και ε, χάσμα, ανισότητα ανάμεσα στα φύλλα. Αυτό να δεικνύει το πρόβλημα και τη σημασία του να ε, προωθήσουμε την ισότητα. Όσον αφορά το συντονισμό των ταμείων, κατανοήσαμε πιο ε, συγκεκριμένα ποιες θα είναι οι ωφέλειες Τώρα έχουμε και το στρατηγικό όργανο το οποίο ε, προσθέτει πλέον χρηματοδότηση πέρα από τα παραδοσιακά μέσα χρηματοδότησης το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. και αυτό είναι κάτι που πρέπει επίσης να δούμε. Κατά δεύτερον, ε, πόσο κινητοποιεί όλο αυτό την ε, δράση σε εθνικό επίπεδο Υπάρχει, έχει αντίκτυπο στο να αλλάξουν συμπεριφορέ στα κράτη-μέλη. Μεμονωμένα, το τρίτο σημείο που θέλω να θίξω και που με, μου προξένησε τον ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπατε για τη χρηματοδότηση με τις χώρες εταίρους σε, άλλους, ε, σε άλλες περιοχές. Με ενδιαφέρει πολύ η Ανατολική Ευρώπη, αλλά αυτό έχει σχέση και με την ε, ε, προσφυγική κρίση για την ενδονάμωση των ε, γυναικών στις περιοχές από όπου ε, προέρχονται οι πρόσφυγες. Τέλος, θίγει και ένα θέμα που έθιξαν και οι ομιλητές, ότι δεν θέλουμε δράση μόνο στη θεωρία. Και θα ήθελα να μάθω αν έχετε κάποια άποψη σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία στην ε, εφαρμογή, πώς θα είναι τα πράγματα τότε και ποια θα είναι η δράση που θα αναλάβετε για να μπορέσετε να τα εφαρμόσετε τελικά όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στις ε, δύο ομιλήτριες, ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας για ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όταν μιλάμε για τον οριζόντιο χαρακτήρα, το gender mainstreaming ή για τις εξειδικευμένε πολιτικές που αφορούν τις γυναίκες. Γιατί το λέω αυτό. Διότι σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, του 2004 νομίζω, στα διαθροτικά ταμεία, είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε εστιασμένες δράσεις και στο ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Κοινωνικό Ταμείο, εστιασμένες δράσεις για τις γυναίκες. Από τη στιγμή λοιπόν που εισαγάγουμε εδώ την αρχή της, του οριζόντιου χαρακτήρα που είναι θετική. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή το θέμα της των δύο φύλων σε κάθε μία από τις δράσεις μας. Αυτό σημαίνει όμως ότι είναι ασύμβατο με εστιασμένα προγράμματα στις γυναίκες. Και δεν μπορεί να πάρθουν κάποια μέτρα που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες γυναικών. Είναι ένα θέμα που το συζήτησα με διάφορες οργανώσεις γυναικών, από τον τομέα της έρευνας, από τον κοινωνικό τομέα, αλλά και του το, τομέα της υπαίθρου μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτή τη στιγμή ε, η, εντύπωση, η εντύπωσή μου, αυτό που ακούω, είναι ότι πρέπει να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα ε, εστιασμένων προγραμμάτων για γυναίκες. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Και εγώ ίδια δεν έχω καταλήξει. Αφενός ε, το gender mainstreaming είναι αυτό που εγγυάται ότι θα υπάρχει η προοπτική ισότητα των δύο φύλων σε όλε τι πολιτικέ. Ταυτόχρονα όμω ε, αυτό χρησιμοποιείται ω δικαιολογία για να μην γίνουν κάποιε συγκεκριμένε ε, παρεμβάσει. Σε σχέση με το, αυτό που είπε η κυρία Μπάνιαν προηγουμένω, ότι πρέπει να συνοδεύεται το gender mainstreaming από μια παρακολούθηση, ε, μια εποπτεία, για να είμαστε βέβαιοι ότι οι στόχοι αυτοί επιτυχάνονται. Και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και επ' αυτού. Ε, σας δίνω το λόγο ευθύς αμέσως για να απαντήσετε. Thank you. That's a lot of, um... Ευχαριστώ. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι... Με συγχωρείτε. Πρώτα να σας πω ότι... Ε, Κάτι που μας δείχνει η έρευνα ως προς το μισθολογικό χάσμα και το χάσμα στις δεξιότητες είναι η παροχή φροντίδας ε, για τα παιδιά. Αυτό είναι ένα ζωτικό θέμα και γίνεται κάποια έρευνα για το γεγονός ότι αν επενδύσουμε στην ε, φροντίδα των παιδιών, τότε δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερο εισόδημα στις εθνικές κυβερνήσεις, περισσότερο κέρδος από ό,τι αν επενδύσουμε π.χ. Ε, στον ε, κατασκευαστικό κλάδο. Και το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι η φροντίδα των παιδιών είναι κομμάτι των υποδομών, θέλετε κομμάτι των υποδομών. Είναι το ίδιο πράγμα όπως είναι και η οδοποιία, όπως οι μεταφορές, γιατί είναι ένα μέσο δημιουργίας θέσεων εργασίας και απασχόλησης, σταθερής απασχόλησης. Άρα θεωρώ ότι είναι κάτι που θα ε, έκανε πολύ μεγάλη διαφορά ώστε να αξιοποιήσουν οι γυναίκες τις δεξιότητές τους, αλλά παράλληλα να αντιμετωπίσουν και το θέμα της ε, ανισότητας ε, στη μισθοδοσία Κάτι που σχετίζεται φυσικά με την φροντίδα των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων παράλληλα. Άλλο θέμα και αυτό. Όλα αυτά επηρεάζουν το συνταξιδοτικό χάσμα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί γιατί θα ήταν χρήσιμο να δούμε λεπτομερώς, να μελετήσουμε παραδείγματα όπου σε χώρες που είναι πιο προσβάσιμη η φροντίδα των παιδιών ε, στην προσχολική ηλικία όπως στην Σκανδιναβία όπου είναι πολύ ψηλής ποιότητας αυτές οι παροχές ε, και δωρεάν τότε είναι πολύ χαμηλότερο και το μισθολογικό χάσμα. Αυτό αφορά βέβαια και το μισθολογικό θέμα, αλλά και το, την ανισότητα στα, στις, στα προσόντα, στις δεξιότητες. Το να αξιολογήσουμε κάποια προγράμματα για να δούμε πώς λειτουργούν, και αυτό είναι κάτι σημαντικό, να δούμε τα συγκεκριμένα μέτρα που αποφέρουν τις μεγαλύτερες ε, βελτιώσεις ώστε να έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες από τα προγράμματα για να υπάρχει και μέτρηση στη συνέχεια, να, υπάρχουν, να είναι και μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Έχω διαχειριστεί και εγώ ένα πρόγραμμα και ξέρω ότι όλη η χρηματοδότηση και όλες οι απαιτήσει ε, αποτελούν ένα κίνητρο για να επιτύχει το, το πρόγραμμα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενσωματώσουμε και την πτυχή του φίλου, το οποίο και αυτό θα αποτελούσε ένα κίνητρο. Πρέπει όμως όλο αυτό να ε, τελεί υπό παρακολούθηση και να εφαρμοστεί στην πράξη. Να δούμε τώρα πώς η εθνική δράση σχετίζεται με την Ευρώπη και να δούμε πώς είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί ο δείκτης ισότητας ε, που ήταν ε, πολύ χαμηλός ανάγκασε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αντιμετωπίσει το θέμα. Ήταν θέμα φήμης, ιστεροφημίας θα έλεγα. Άρα και τέτοιου είδους ε, παράγοντες βοηθούν και παράλληλα συγκεκριμένες δραστηριότητες για τις γυναίκες και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε θέματα σε συγκεκριμένους τομείς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χρηματοδοτούμε απλά κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη ισότητα, αλλά ότι θα κρατήσει κάποιες γυναίκες σε συγκεκριμένους κλάδους εργασιακούς να υπάρχουν πολύ προσεκτικές μετρήσεις ώστε να έχουμε μετρήσιμη βελτίωση. Όταν υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών, τότε προφανώς πρέπει να αναπτυχθούν οι δεξιότητες τους. Θα να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, θέματα και να δημιουργήσουμε, ε, να βρούμε στοιχεία που θα οδηγήσουν σε, στη βελτίωση της κατάστασης. Όσον αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, και αυτό πολύ μας ενδιαφέρει. Πρέπει παράλληλα επίσης να αξιολογήσουμε πόσο αποδοτικό είναι αυτό όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε στρατηγικές θέσεις στις επιχειρήσεις, γιατί κάποιες, ε, κάποια στοιχεία που έχουμε από την Νορβηγία δείχνουν ότι <coughs> υπάρχουν πολύ περισσότερε απαιτήσει από τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια και ότι αυτό δεν έχει δημιουργήσει αλλαγέ ουσιαστικά στην ανισότητα των, τη μισθολογική ανισότητα. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν είναι η αποτελεσματικότητα και η επίδραση που έχει αυτό στα διοικητικά συμβούλια αν απλώς προωθεί συγκεκριμένες γυναίκες ε, μπορεί να είναι καλό γενικά ε, για την φήμη μας αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο αποδοτικό. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω από τα όσα είπε η βουλευτήνα του ΕΛΚ. Ε, αυτά τα τρία σημεία μας οδηγούν σε ένα ιδανικό κόσμο. Ε, η Ιταλία, ε, όπως σας είπα, Ταλίδα και ακριβώς βλέπω τα πράγματα μέσα από το τι γίνεται χώρα μου και έχουμε και τις ευρωπαϊκές στατιστικές, άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά της απασχόλησης. Είναι το θέμα της μισθολογικής ισότητας. Αυτό είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή που κατοχυρώθηκε πρώτη φορά το 19. Ε, έχει γίνει μια διαδρομή μισού αιώνα από τότε, αλλά έχουμε το 16% του μισθολογικού χάσματο. Και έχουμε και τα στερεότυπα επομένω να αντιμετωπίσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα από την εμπειρία μου και πανεπιστημιακή αλλά και μέσα από καταρτήσεις, εκπαιδεύσεις ε, θεωρώ ότι η υπόθεση της ισότητα των ευκαιριών είναι μια προτεραιότητα για εκπαίδευση και κατάρτιση. Όμως ακόμα από τα προγράμματα χρηματοδότησης ε, δεν έχει πλαισιωθεί. Αυτό έχω καταλάβει. Επομένω, αν εκεί κάνουμε το πρόοδο, θα κάνουμε τη διαφορά. Να ποια είναι η ισότιμη δημοκρατία. È un processo lunghissimo che tantissimo tempo, Μια δημοκρατία, μια πολιτεία ίσων ευκαιριών. Είναι και θέμα ε, κουλτούρα. Συγκεκριμένε δράσει χρειάζονται. Αυτό ε, το οποίο ανέφερε προηγουμένω η πρώτη ομιλήτρια χρειάζεται ισότητα ενώπιον του δικαίου αλλά να μην ξεχνούμε ότι χρειάζεται και το mainstreaming επομένως συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της κοινωνίας θα πρέπει να αναλυθούν και να πλαισιωθούν αλλιώς οι νόμοι μένουν νεκρό έχουμε τις ποσοστώσεις, τις ροζ ποσοστώσεις όπως τις λέμε αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά υπάρχουν σε διάφορες δημοκρατίες. Σε Νορβηγία, σε... Ε, ε, Σουηδία, αλλά δεν υπάρχει όμως στην πράξη η εκπροσώπηση. Το βλέπουμε αυτό να ισχύει ακόμα και μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Άρα χρειάζεται τέτοια πολιτική για το mainstream και για την ισότητα ευκαιριών που θα πρέπει να πιάσει τόπο, να ριζώσει και έτσι θα οδηγηθούμε σε πραγματική ισότητα ευκαιριών. Είναι κάτι σαν πολιτιστική επανάσταση που πρέπει να γίνει. Είδατε τι έγινε πρόσφατα στην ε, Πολωνία. Δεν είναι επομένως κάτι το κατακτημένο, το κεκτημένο η υπόθεση των δικαιωμάτων της γυναίκας. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει κανείς να δίνει κάθε μέρα αγώνα. Είναι συνεχές το ζήτημα. Δεν είναι καν κάτι που εντοπίζεται μέσα στην ε, οικονομική κρίση. Δεν είναι ένα θέμα επίσης, ένα υποθέμα το οποίο ακριβώς αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της κρίσης. Είναι το θέμα η ισότητα ευκαιριών. Αν ποια είναι η πραγματική δημοκρατία ίση συμμετοχή. Έχουμε και τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Και επίση αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο τώρα στην Ιταλία σε εκπαίδευση και παιδεία. Τώρα, τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά ταμεία τι γίνεται με την άμεση και την έμεση υποστήριξη από οικονομικής πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουν τη διαφορά. Καλύπτουν τις εταιρείε και τα νομικά πρόσωπα. Εξαρτάται βέβαια και από το τι κουλτούρα, τι πνεύμα επικρατεί σε κάθε χώρα. Θα πρέπει να αναδεικνύονται και να υποστηρίζονται οι σωστές πρακτικές. Και χρειάζεται επίσης συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών και να διαδίδονται αυτές οι καλές πολιτικές. Οπότε να επιφέρουμε βελτιώσεις με δράσεις. Και έτσι θα φτάσουμε στην αλλαγή, στη διαφορά. Να, πώς θα βοηθήσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης. Δύσκολη και αυτή η φάση. Και δεν θα πρέπει επομένως να χαθεί το τρένο όπως είπε η Ευρωβουλευτής από την Τσεχία. Να δούμε ποια είναι τα πιο δόκιμα προγράμματα και έργα. Και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και τις δύο εισηγήτριες για τα όσα μας είπαν στην αρχή, αλλά και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους θέσαμε. Σίγουρα όλα αυτά θα μας βοηθήσουν στο έργο μας και συγκεκριμένα στην έκθεση αυτή. Τώρα έχουμε το δεύτερο πάνελ. Έχουμε άλλους δύο καλεσμένους. Παρακαλώ να έρθουν για να συνεχίσουμε ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε λίγο καθυστερήσει σε σχέση με το πρόγραμμα. Vamos a comenzar Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το δεύτερο πάνελ. Όπως σας είπα, επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω, θα ζητήσω και από τους δύο ομιλητέ ε, να προσπαθήσουν να μην ξεπεράσουν τα 10 λεπτά ε, για να έχουμε χρόνο στη συνέχεια να ακούσουμε και τις ε, και τους ευρωβουλευτές Λοιπόν, η κυρία Μανουέλα Σάμεκ Λουντοβίτσι από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας από την Ιταλία ειδική στα ζητήματα στους των δύο φύλων και διατροτικών ταμείων. Παρακαλώ. Okay. Ε, yes. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Είναι μια μελέτη πάνω στην οποία ακόμα εργαζόμαστε, άρα τα σχόλια θα είναι πολύ χρήσιμα για μας, για να προχωρήσουμε. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να αξιολογήσουμε τις, ε, τα στοιχεία για το πώς το gender mainstreaming εφαρμόζεται ε, στις, ε, στην κατανομή των ευρωπαϊκών ταμείων, με εστίαση κυρίως τη χρηματοδότηση για την ε, φροντίδα των παιδιών, υπό τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία η ένταξη του, της πτυχής του φίλου στον ΕΣΔΟ 2020, gender mainstreaming στα προγράμματα REC και κυρίως ο στόχος και την ισότητα των φίλων ε, στο πρόγραμμα DAFNE και κυρίως στις χώρες που βλέπετε, την Κροτία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σουηδία και τον Εμένο Βασίλειο βασίσαμε τη μελέτη κυρίως σε μία ανάλυση ε, χρηματοπιστωτικών δομένων και σχετική τεκμηρίωση προκηρύξεις, χρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσπαθήσαμε να δούμε τι έχει γίνει μεταξύ 2014 και ε, Σεπτεμβρίου 2016. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι, ότι η κατάρτιση προπολογισμού σύμφωνα με το φύλλο είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για το gender mainstreaming, γιατί χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις. Το gender budgeting, λοιπόν, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την ενσωμάτωση της πτυχής ε, του φίλου. Το gender budgeting δεν εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα τα χρηματοδοτούμενα. Και επίσης το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο του 2014-2020 περιλαμβάνει μια γενική ανακοίνωση, μια κοινή ανακοίνωση για τη σημασία του gender mainstreaming και την ανάγκη της χρήσης του gender mainstreaming στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όμω, η ισότητα των φύλων δεν είναι ανάμεσα στου βασικού στόχου και γι' αυτό υπάρχουν πολύ λίγα ταμεία που αφορούν την ισότητα και δεν υπάρχει αρκετή προσοχή για το πώς τα άλλα ταμεία εφαρμόζουν το gender mainstreaming. Βλέποντας ε, και την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση του πολιτικού συνδεμοσιονομικού πλαισίου που προτείνονται κάποιες αλλαγές και μετατροπές ε, στην κατανομή του προπολογισμού δεν υπάρχει αρκετή προσοχή πάλι σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων και το gender mainstreaming. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι με το gender mainstreaming, την ενσωμάτωση της διάθεσης του φύλου, είναι εύκολο να πούμε σε μια γενική διατύπωση ότι θα το λάβουμε υπόψη σε όλα τα προγράμματα, το gender mainstreaming, αλλά όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος, ε, πόρη για την ισότητα των φύλων, τότε είναι πολύ δύσκολο το gender mainstreaming να εφαρμοστεί επιτυχώς. Και υπάρχουν παράλληλα, υπάρχει πολύ λίγη πληροφόρηση οι πληροφορίες που έχουμε για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση για την εφαρμογή αυτών των ε, ταμείων δεν ξεχωρίζει τα ταμεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη ε, της ισότητας των φύλων σε σχέση με άλλα ταμεία που δεν είχαν συγκεκριμένους στόχους. Τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία για την πολιτική συνοχής, αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου του προπολογισμού για το 2014 το 2020 και είναι και τα πιο σημαντικά από πλευρά πόρων για την ε, υποστήριξη της ε, πολιτικής ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι κανονισμοί κάνουν αναφορά στο gender mainstreaming. Υπάρχει ε, συγκεκριμένη διατύπωση για το πώς πρέπει τα ταμεία να υποστηρίζουν την εφαρμογή του gender mainstreaming. Είναι μια αιρεσιμότητα ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όργανα αρμόδια για την ισότητα, ότι πρέπει να γίνεται μελέτη δικτύπου κτλ. Ότι θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση των δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δείκτες που αφορούν πάλι την ισότητα των φύλων. Όμως δεν υπάρχει δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι επιλεγμένοι πόροι για την ισότητα. Περνάει σε δεύτερη μοίρα, επομένως, προς όφελος άλλων θεμάτων. Άρα το gender mainstreaming δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί, ειδικά σε ταμεία που δεν περιλαμβάνουν αποκλειστικά ε, άτομα όπως ε, τα ταμεία για την ανάπτυξη πέθρου, τη γεωργία κτλ. Σε αυτά τα ταμεία οι αρχές διαχείρισης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει για την προώθηση της ισότητας σε, αυτές, σε αυτούς τους τομείς της πολιτικής. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. και στα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων. Άλλες πτυχές αναφέρονται στα, αφορούν τα κοινωνικά ταμεία, στο κοινωνικό ταμείο, η ισορροπία ανάμεσα στην ζωή και την εργασία, στην προσωπική ζωή και την εργασία, παραδείγματο χάρη, και περιλαμβάνονται και στον θεματικό στόχο 9, που θα πρέπει, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να υποστηριχθεί και η φροντίδα των παιδιών. Από τις επιτροπές φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν Υπάρχουν 5 ε, δισεκατομμύρια 850 ε, εκατομμύρια και 25 εκατομμύρια άλλο ταμείο για να υποστηρίξουν ε, συγκεκριμένες δομές και υποδομές ε, για τα παιδιά. Όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας και τη φροντίδα των παιδιών, οι πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες έχουν να κάνουν με την περίοδο 2014-2020. Υπάρχουν 1,6 ε, εκατομμύρια στο πρόγραμμα ESF για την ισότητα των φύλων Κάτι που κάνει και πάλι αναφορά στην ισορροπία μέσα σε προσωπική ζωή και εργασίε. Αυτό επιλέχθηκε από 12 κράτη-μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, τότε τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιλέξουν πού θα επενδύσουν. Approach of concentrating resources on the 12 κράτη-μέλη, λοιπόν, έχουν επιλέξει αυτούς το ως προτεραιότητα και θα ε, εξοπλίσουν και το στρατηγικό ταμείο ε, το, το στρατηγικό επενδύσεων ε, στο θέμα της φροντίδας των παιδιών. Δεν γνωρίζουμε ακόμα Ε, πώς θα εφαρμοστεί αυτό, αυτό όμω αναμένεται και ε, από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν έχουμε την έκθεση αιτήσεις εφαρμογή. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πώς τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες επενδύουν για αυτές τις προτεραιότητες. Κοιτάζοντα τα επιχειρησιακά προγράμματα των έξι κρατών μελών που θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο, αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσει και στρατηγικέ στα επιχειρησιακά προγράμματα. Στην Σουηδία δεν χρειάζεται να αξιοποιήσουν τα αντιρρητικά ταμεία για να υποστηρίξουν ε, τι υπηρεσίε για τα παιδιά, γιατί η Σουηδία ήδη είναι μία από τις χώρες, από τις καλύτερες χώρες σε αυτό το τομέα. Έχουν επενδύσει τα μέγιστα σε εθνικό επίπεδο. Άρα το στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων θα υποστηρίξει κυρίως ε, το gender mainstreaming, τη δημιουργία δομών που θα βοηθήσουν ε, τα Υπουργεία στην ε, προώθηση του gender mainstreaming. Στη Γερμανία Υπάρχει κάτι παρόμοιο. Έχουν και οι δύο επενδύσει σε υπηρεσίε για τη φροντίδα των παιδιών, γιατί είναι από τι χώρε που έχουν επιλέξει την προτεραιότητα ε, επένδυση που ανέφερα πριν. Αλλά από το 2009 έχουν δημιουργήσει αυτή την υπηρεσία ισότητα των φύλων που παρέχει τεχνική ε, βοήθεια τόσο στα Υπουργεία όσο και σε ε, διαχειριστές προγραμμάτων για την αξιοποίηση του gender mainstream στο πλαίσιο των διευθυντικών ταμείων. Στην Ιταλία, επισήμως, η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται στην εταιρική συμφωνία συμφωνία εταιρική σχέση και υπάρχει και παρέμβαση σε κάποιους ε, τομείς για την ε, φροντίδα των παιδιών, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ESF και στον τομέα της ισορροπίας ζωής, ε, προσωπικής ζωής και εργασίας. Αλλά στο πλαίσιο του ERDF υπάρχουν λίγες αναφορές σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει. Η Πολωνία και η Κροατία είναι οι δύο χώρες που επενδύουν περισσότερο στα επιχειρησικά τους προγράμματα για τις υπηρεσίε για τα παιδιά και για τις υποδομές, σχετικές υποδομές. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυψης για τη φροντίδα των παιδιών και για να αυξήσουν το ποσοστό κάλυψης για να επιτύχουν και το στόχο της Βαρκελόνης θα επενδύσουν και από το ESF και από το ERDF για την ανάπτυξη υπηρεσίων ε, σε κοινωνικό επίπεδο και πρωτοβάθμιες υγείας επίσης. Ειδικά στην Πολωνία, σε πολλά περιφερειακά προγράμματα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τον αριθμό των παιδιών που θα θελήσουν να εντάξουν σε αυτά τα προγράμματα και σε υποδομές αντίστοιχες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα διευθυντικά ταμεία θα στηρίξουν την ε, φροντίδα των παιδιών και την ισορροπία ζωής ε, εργασίας, κάποια επιχειρηστικά προγράμματα εστιάζουν ε, σε μονογονεϊκές οικογένειες, έξι επιχειρησιακά προγράμματα, ε, υποστηρίζουν ε, ευέλικτες πρακτικές εργασίας σε εταιρείες, και κάποιοι επίσης προγράμματα ε, υποστηρίζουν τη φροντίδα των παιδιών, χρησιμοποιώντας άλλα ταμεία. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών. Στον ορίζοντα τώρα περνάμε. Υπόθηκε κάτι πριν, άρα δεν θα, το... δεν θα τους στόχους. Στον ορίζοντα υπάρχει μία ισχυρή δέσμευση ως προς το gender mainstreaming και υπάρχει συγκεκριμένο ταμείο, το Jerry fan στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά α, το ταμείο για τη διάσταση του φύλου, Αν δούμε όμω πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό το 2014-2015, βλέπουμε όλα τα προγράμματα που υποστηρίχθηκαν. Από τα 10.000 και περισσότερα προγράμματα που υποστηρίχθηκαν από το ορίζοντα 2020, μόνο 71 είτε άμεσα είτε έμεσα ε, αγγίζουν θέματα ισότητας φύλων. Πολύ μικρό το ποσοστό λοιπόν. Βλέπετε στη διαφάνεια υπό ποιο πυλώνα βρίσκονται αυτά τα προγράμματα. Στην τελική έκθεση υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα. Όσον αφορά ε, το Ταμείο Τζέρι, που αφορά αποκλειστικά προγράμματα ισότητας φίλων υποστηρίζει οργανώσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων, την αξιολόγηση πρωτοβουλειών, μεθοδολογιών, την, ε, την αξιολόγηση του αντικτύπου, έρευνα, καινοτομία και καινοτόμες προσεγγίσεις στο θέμα της ισότητας των φύλων. Έχουν γίνει προκηρύξεις για 19 εκατομμύρια ευρώ και 9 προγράμματα έλαβαν χρηματοδότηση και τα πιο πολλά από αυτά τα προγράμματα υποστηρίζουν ε, ερευνητικούς φορείς. Βλέποντα τις έξι χώρε, ε, αυτό που προκύπτει είναι ότι κυρίως η Γερμανία από τον Τζέρι και η Ιταλία στη συνέχεια είναι σε ηγετική θέση. Η Γερμανία είχε, είχε τρία προγράμματα από τα νέα προγράμματα και η Ιταλία είχε ένα από τα νέα προγράμματα. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα προγράμματα, 71 προγράμματα του ορίζοντα που αφορούσαν το ίδιο θέμα, διεξάχθηκαν κυρίως από ε, βρετανικούς οργανισμούς. 33 προγράμματα συνολικά. Όσον αφορά το ταμείο αυτό, το Τζέρι, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ε, μία συγκέντρωση υπογραφών από ακαδημαϊκούς και ερευνητές γιατί υπάρχει κίνδυνος αν ε, δούμε το πεδίο εφαρμογής τα επόμενα δύο χρόνια και τον προϋπολογισμό για τον ορίζοντα, ο κίνδυνος είναι ότι το Τζέρι δεν θα είναι ανεξάρτητο το χρηματοδοτικό ε, μέσο, αλλά θα συμπεριληφθεί ε, στην ε, χρηματοδοτική γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας. Και έτσι θα χάσει την ισχύ του και την δυναμικότητά του. Άρα υπάρχει μια συλλογή υπογραφών για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Τώρα, το πρόγραμμα REC. Υπάρχουν δύο στόχοι ισότητας ε, μεταξύ των φύλων. τον DAFNE που προωθεί την ε, ισότητα μεταξύ των φύλων και τον gender mainstreaming και το άλλο είναι DAFNE που θέλει να αντιμετωπίσει τη βία εναντία στις γυναίκες και στα παιδιά. Αυτοί οι δύο στόχοι αφορούν το 35% του συνολικού προπολογισμού του ΡΕΚ και αν δούμε τι έχει γίνει μέχρι, το, μέχρι μεταξύ 2014 και Σεπτέμβριο του 2016 προκύπτει ότι ότι από τα τις 70 χρηματοδοτήσεις και τα 65 προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν υπό το ΡΕΚ, μόνο τα 7 με τα 46 προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί ε, μόνο τόσα έχουν χρηματοδοτηθεί που έχουν ως στόχο την ισότητα των φύλων. Και τα πιο πολλά έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση με τις γυναίκες. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Τα επιλεγμένα προγράμματα, ποιες προτεραιότητες έθεσαν για το Δάφνη το 39% των πόρων απορροφήθηκαν για την καταπολέμηση της ε, βίας. Την καταπολέμηση του εγκλήματος, την καταπολέμηση και την... Ε, το θέματα που φορούν την κλίτερη δεκτόμη κτλ. Μεγαλύτερη χρηματοδότηση πήγε στην οικονομική ε, ανεξαρτησία των γυναικών και την εξορρόπηση και την προώθηση των ορθών πρακτικών. Για να ε, καταλήξουμε και θα ολοκληρώσω εδώ. Ξεκάθαρη στρατηγική για την ισότητα, πέρα από αυτά που ε, λέγονται, δεν προκύπτει από το πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχει χαμηλή υποστήριξη για ανάληψη δράσης που να στοχεύει στην ισότητα των φύλων. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πόροι που κατανέμονται συγκεκριμένα για τέτοιους στόχους, δίκτες, μελέτες αξιολόγησης και εργαλεία ε, της προπολογισμού που είναι πολύ χρήσιμα για το gender mainstreaming. Όλα αυτά πολύ σπάνια λαμβάνονται υπόψη και υιοθετούνται στην ε, εφαρμογή πολιτικής ε, και στην αξιολόγηση βέβαια της κατανομής του προπολογισμού και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι άλλο που προκύπτει είναι ότι συνήθως τα θέματα φύλων αντιμετωπίζονται περισσότερο σε ήπιες, τομεί τομείς πολιτικής, κοινωνικές πολιτικής, τέτοιου είδους και πολύ λιγότερο σε σκληρούς τομείς ε, πολιτικής, βαρύ, ε, σημαίνοντες τομείς, όπως είναι οι υποδομές που αποτελούν και το μεγαλύτερο ε, κομμάτι των χρηματοδοτικών πόρων. Οι προτάσει είναι να υπάρξει ισχυρότερη δέσμευση για την ισότητα των φύλων και την ε, συμπερίληψη της διάσταση του φύλου και να είναι πιο δεσμευτική προσέγγιση. Θα πρέπει συγκεκριμένα ποσά να ε, κατανέμονται, ε, να πιστώνονται για τέτοιες δράσεις που υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων. Ε, η κατάρτιση προπολογισμού συγκεκριμένα για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να ε, υπάρξει επίση και να υπάρξει δέσμευση για στόχους να υπάρξουν ε, και να υπάρξει κατάρτιση δικτών, να υπάρξει και ε, κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων που προετοιμάζουν τον προϋπολογισμό ώστε να γνωρίζουν τι είναι το gender mainstreaming και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Yo, yo eh, mm, Συγγνώμη που σα έκοψα, αλλά ξέρετε πρέπει να συμμετάσχουν όλοι στη συζήτηση ε, και διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε. Ούτω ή άλλω δεν θα μπορέσουμε δηλαδή, να έχουμε συζήτηση από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριο Σκάνα τώρα, υπεύθυνο ε, για ζητήματα κοινωνική εκπαίδευση και οικογενειακή πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Εισηγήτρια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση εκ μέρους ε, του οργανισμού μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι, είναι πραγματικά τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι και ο μόνος άντρας εδώ στο πάνελ. Θα εκπροσωπήσω λοιπόν το ανδρικό φύλλο. Ε, θα προσπαθήσω να μιλήσω λιγότερο από τα 10 λεπτά που μου αναλογούν για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφο. Εκλήθην εδώ για να μιλήσω για τα ζητήματα των πολιτικών, των ταμείων και να κάνω μια εισαγωγή ε, σε ό,τι αφορά ε, τα προγράμματα για το gender mainstreaming και την επίπτωσή τους στην Τσεχία, τον αντίκτυπό της στην Τσεχία και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε. Θα είμαι εξαιρετικά συγκεκριμένος. Ζητώ συγγνώμη ε, για όσους δεν αρέσουν οι εικόνες εδώ και οι ζωγραφιές. Πρέπει να πω ότι μόλις ε, είδα αυτή την εικόνα ε, εμένα μου άρεσε αμέσως. Είναι ένας καλός τρόπος για να μιλήσουμε για την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων ακόμα και αν έχει έτσι ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Λοιπόν, τα ζητήματα που θα αναφέρω όμως είναι σοβαρά και ελπίζω να τα ακούσετε προσεκτικά. Η Τσεχία έχει εμπειρία στον τομέα αυτών παρότι αυτή η εμπειρία δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και όταν ήμασταν στο, πρόγραμμα FAIR, υπήρχαν κάποια εστιασμένα προγράμματα για ισορροπία μεταξύ ε, ζωής, ε, πραγματική ζωής, ε, για την πρόσβαση στην απασχόληση, για τις μειονεκτούσες ομάδες, για τις γυναίκες μετά το, τη μητρική άδεια, την άδεια μητρότητα, έχουν επενδυθεί σημαντικά ποσά προ την κατεύθυνση αυτή. Όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισαμε να χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα πλαίσια, τα οποία είναι γνωστά σε όλου. Αρχίσαμε να ε, βρίσκουμε επενδύσει από εκεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξη ε, των ανθρωπίνων πόρων και τη απασχόληση και υπάρχει μια ειδικά εστιασμένη ε, δράση για την ε, ευξήση ευκαιρία για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Ε, αν θέλουμε λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα οικονομικό πλαίσιο, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, το, κατά την κάθε προγραμματική περίοδο στην Τσεχία, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε μια συγκεκριμένη πτυχή του ζητήματος μεταξύ του ζητήματο τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Να ξέρουμε δηλαδή επακριβώ ποια ποσά διαθέτουμε πού. Από την άλλη, η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα οριζόντιο κριτήριο το οποίο έχει θέση σε κάθε άλλο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν τα πραγματικά ποσά τα παιδιά διατίθενται για το ζήτημα αυτό είναι πιο σημαντικά, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το κάθε άλλο πρόγραμμα ε, το οποίο ε, χρηματοδοτούμε πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν δημιουργεί διακρίσεις κατά των γυναικών και ότι λαμβάνει υπόψη την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία για την περίοδο 2004-2006. Μιλάμε για περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Σε αυτή την περίοδο εμείς συμμετείχαμε στο CIP Equal. Τώρα έχουμε την περίοδο 2007-2013 βέβαια ε, υπήρξε ένα σχέδιο για την απασχόληση και μια ιδιαίτερη πτυχή που αφορούσε τις ίσες ευκαιρίες ε, ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Δύο εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν, ή ε, μάλλον 42 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν. Και χρησιμοποιήθηκε ποικιλό τρόπο αυτό το πρόγραμμα και τώρα για την παρούσα ε, προγραμματική περίοδο. Έχουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα ε, για την απασχόληση. Υπάρχει ε, εδώ ένας συγκεκριμένος στόχος να μειωθεί η απόκληση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. αυτό που διαπιστώνουμε εδώ με ενδιαφέρον είναι ότι είναι πολύ υψηλότερα τα ποσά που διατίθεται. 244 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε βεβαίως πόσα από αυτά θα απορροφηθούν, αλλά αυτό είναι το ποσό που διατίθεται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει αυτό το φαινόμενο ε, να μην αποτελεί πλέον θέμα προτεραιότητας αυτό, αυτός ο στόχος σε κάποια Δεν ισχύει όμως αυτό στην Τσεχία καθόλου. Είναι το τρίτο πιο χρηματοδοτούμενο θέμα ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ιδέες ε, για τα διάφορα project δεν βασίζονται μόνο σε στεγνές εκθέσεις. Έχω και εγώ προσωπική εμπειρία. Έχω συμμετάσχει σε κάποια από τα project αυτά. Συνεργάστηκα με την ομάδα εστίασης γυναικών, εστίασης μάλλον στις γυναίκες που επιτρέφουν, επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ε, άδεια μητρότητας. Κάποιες από αυτές είναι στην ανεργία, κάποιες άλλες ομάδες γυναικών ε, στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού. Συμμετείχα στο πρόγραμμα ήδη από το 2004-2006. Τότε υπήρχε ένα μεγάλο project για την ισότητα στην Βυσότσινα. Η Βυσότσινα είναι μια περιφέρεια ε, αυτοδιαχειριζόμενη ε, στη Τσεχία και ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους έφτασε, είχε αντίκτυπο αυτό το πρόγραμμα, ήταν πάνω από χίλιες γυναίκες. Ε, και βεβαίως από αυτά τα προγράμματα έχουμε ένα feedback. Ε, τέθηκαν κάποια ζητήματα ε, για τα κοινά, για τα commons. Όλοι ζητούν συγκεκριμένες συστάσεις για, για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας προς όφελος ε, των γυναικών για τη βελτίωση, δηλαδή ε, την θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό που έχουμε κάνει στα πλαίσια των project αυτών είναι ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε στις γυναίκες ε, μια χείρα βοηθείας. Μετά από μια περίοδο που δεν συμμετείχαμε, ε, που οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στην αγορά εργασίας, που είχαν αποσυρθεί για διάφορους λόγους. μου ζητήθηκε να μην, να μην είμαι γενικόλογος και αυτό θέλω να το σεβαστώ αλλά αξίζει νομίζω να αναφέρω γιατί κάποια πράγματα δεν λειτουργούν καλά. και γιατί κάποια μέτρα δεν βρίσκουν κοινό, δεν βρίσκουν ανταπόκριση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε η Τσεχία να εφαρμόσει τα προγράμματα ήταν μια προσπάθεια να αποφύγουμε το ιδεολογική, την ιδεολογική προσέγγιση. Το 2004 υπήρχε ένα εγχειρίδιο για το gender mainstreaming, το οποίο μεταφράστηκε στα τσεχικά. Όσοι λοιπόν θέλουν να ξέρουν περισσότερα μπορούν να το πράξουν. Ε, μπορούν να ενημερωθούν, έχουν τις πληροφορίες στη διάθεσή τους. Όμως δεν πρόκειται να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, ας αναρωτηθούμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Εγώ ασχολούμαι με το στρατηγικό πραγματισμό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να βρουν τη θέση τους στον κόσμο να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν με βάση τις δικές τους προτεραιότητες στη ζωή πώς θέλουν να οικοδομήσουν το μέλλον τους, την καριέρα τους, ποιες είναι οι προτεραιότητες τους, πώς τις ιδιαρχούν Και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Δεν θα μιλήσω τώρα για στατιστικά στοιχεία εδώ. Υπάρχουν όμως κάποιοι, κάποιες ενδείξεις που έχουμε του ακούσαμε τις γυναίκες τίθενται κάποια ερωτήματα ε, ποια είναι τα καλύτερα μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν για να, βοηθήσουμε τις γυναίκες να επιστρέψουν στο... στην αγορά εργασίας όταν έχουν αποσυρθεί για ένα διάστημα όλα αυτά τα έχω συνοψίσει σε τρία συγκεκριμένα σημεία πρώτον θα πρέπει να υποστηρίξουμε την στρατηγική για, την, ε, για τις ευκαιρίες. Πρέπει να νιώθουν οι γυναίκες ότι τα μέτρα που προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι προς όφελός τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες μαζί και οι δύο θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο, ε, να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στις γυναίκες έτσι ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι ίδιες, να αυξηθεί δηλαδή η αυτοεκτίμησή τους. Όταν μιλά, μιλήσαμε στις γυναίκες στην περιοχή της Βυσότσινα, κάποιες από αυτές δεν είχαν δουλέψει 8-9 χρόνια. Δεν ήξεραν πώ να επιστρέψουν στην αγορά εργασία. Κάποιες είπαν, ακούστε, έχω να δουλέψω τόσα χρόνια, εάν τώρα αρχίσω ε, να δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ, να γεμίζω τα ράφια, ε, για μένα καλό είναι. Δημιουργήσαμε λοιπόν ομάδε ε, και αρχίσαμε να μιλάμε για τι αδυναμίε τη κάθε γυναίκα αλλά και τα ισχυρά τη σημεία, τα πλεονεκτήματά του και κάποιοι κάποιες γυναίκες μόνες τους έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το να δουλεύουν σε ένα σούπερ μάρκετ ε, δεν είναι το πλέον ενδεδειγμένο σε σχέση με τα προσόντα τους, σε σχέση με τις δυνατότητές τους, ε, το, τα, τα ταλέντα τους ε, και αποφάσισαν να στοχεύσουν λίγο πιο ψηλά, να δουλέψουν σε μια γραμματεία. Αποφάσισαμε λοιπόν να βελτιώσουμε ε, την ευαισθητοποίηση των γυναικών αλλά και των εργοδοτών. Πολλές συχνά οι εργοδότες ε, υποβάλλουν τις γυναίκες στη διακριτική μεταχείριση. Πληρώνονται λιγότερο για την ίδια δουλειά. Συχνά ο εργοδότης χρησιμοποιεί την ευκαιρία το, ναι. την ευκαιρία ότι η γυναίκα δεν γνωρίζει πόσο πρέπει να πληρωθεί ε, η οποία δέχεται ένα χαμηλό ποσό. Από εκεί πρέπει να αναπτύξουμε εμείς κάποια εργαλεία υποστηρικτικά για να βοηθήσουμε τις γυναίκες ε, να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να είναι καλύτερες σε μια διαπραγμάτευση ε, για την αμοιβή τους. Αυτός είναι ένας τρόπος ε, για να ελαχιστοποιήσουμε ε, το κενό, το χάσμα αμοιβών. 80 με 100 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη θεωρούν τη μητρότητα ανεξαρτητικά σημαντικό στοιχείο στη ζωή τους. Αλλά είναι μεγάλα και τα ποσοστά των γυναικών που θεωρούν ότι και η καριέρα τους έχει σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε τις γυναίκες ως μητέρες να μην τους πούμε ότι το ένα ή το άλλο έχει μεγαλύτερη σημασία να τους βοηθήσουμε να βρουν την, το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματική του ζωής και βεβαίως χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη για τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία στο σπίτι πρέπει εδώ να είμαστε πιο ενεργοί. Ορισμένε φορές ε, ε, υπάρχει ένας φόβος για το πώς θα μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε η οικογενειακή ζωή και η πραγματική ζωή. Συχνά αυτό οδηγεί σε διαζύγια και συχνά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε περισσότερη δουλειά στον επίπεδο της πρόληψης εδώ. Και βεβαίως υπάρχουν και οι μη επιθυμητές επιπτώσεις των πολιτικών μας. Ορισμένες φορές έχουμε καλή βούληση, έχουμε ε, καλό σκοπό, ε, σκεφτόμαστε πώς θα λειτουργήσει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα εξελίσσονται αλλιώ. Ε, κάνουμε λάθη. δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι, που θέλει οι διακρίσεις στην Ευρώπη να εξαλειφθούν. Όλοι θέλουμε οι πολιτικές μας ε, να πετυχαίνουν το σκοπό τους. Η επίτροπά μας, η κυρία Γιούροβα, έχει πει κάτι σημαντικό επ' αυτού. Είμαι να απαντήσω, είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Two experts, uh, Mr. Skalka. Να ευχαριστήσω τους δύο ε, εισηγητές, τον Σκάλα και τον Λουντοβίτσι. Σκάλα και τον Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι 5 και 5, άρα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε κατευθείαν στο επόμενο σημείο της μερισίας διάταξης, που είναι η παρουσίαση μιας μελέτης από τον κύριο Μασκερίνη, που είναι διευθυντής έρευνας στο, στη μονάδα του Eurofound για την απασχόληση και την αλλαγή για τις ε, προκλήσεις και τις λύσεις ε, στην ισότητα των φύλων. Mr. Mascarini, if you would like, like to start, please. Okay. Thanks, Madame la President. Ladies and gentlemen. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από πλευράς Eurofound να σας ευχαριστήσουμε που μας προσκαλέσατε στο Κοινοβούλιο. Μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα σχετικά με μισθολογική ανισότητα. Πρώτη, για τη διαφορά ε, όσον αφορά την αμοιβή ανδρών και γυναικών, δηλαδή περίπου το 10% είχαμε σαν, ε, σαν διαφορά το 15%. Οπότε πρόκειται για όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες ε, δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην αγορά απασχόληση αλλά και υποχρέσεων δεν έχουν την ευκαιρία να το πράξουν και σε αυτή την παρουσίαση, αλλά επίσης και στην έκθεση που δημοσιοποίησαμε, λέμε για το πώς θα μπορούσε να έρθει αυτή η διαφορά, αυτή η ανισότητα σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο ατόμου. Να δούμε ποιο είναι το κόστος αυτής της ανισότητας για την Ευρώπη. Να δούμε επίσης τι γίνεται με τις πολιτικές, για το ότι χρειάζεται παρέμβαση μια πολιτική για να αρθεί η ανισότητα. Σε ατομικό επίπεδο τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρθεί η ανισότητα για να υπάρξει οικονομική ανεξαρτησία, ούτως ώστε γυναίκες και άντρες να μπορέσουν να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και της οικογένειας τους. Έχουμε βέβαια τις μορφικές μεταβολές έχουμε αυξανόμενη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να υλοποιήσουμε τους στόχους του θεματολογίου ορίστον 2020. Πρόκειται για κάποιες ε, πρωτοβουλίες για την ισότητα, πρόκειται για την δέσμη επενδυτικών μέτρων και πρόκειται και για τον χάρτη πορείας. Για μια καινούρια αρχή, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Παρά την ε, αύξηση οι άντρες απασχολούνται κατά 70,1% και οι γυναίκες μόνο 59,6% παρά την αύξηση των πληθυσμών. Βέβαια υπάρχουν ποικιλίε ανά κράτος μέλος, διαφοροποιήσεις και έχουμε 41,1% στην Ελλάδα και πάνω το 73% στην ε, Σουηδία. Οπότε βέβαια είναι ε, ετερογενές το περιβάλλον στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ανισότητα σε όλα τα κράτη-μέλη και βέβαια η διαφορά ε, είναι άνιση μεταξύ των μελών. 1,5% στη Φιλανδία και 25,6% στην Μάλτα. Πάντω συνολικά διαπιστώνουμε όταν θέλουμε να δούμε τι πάνε να το 10% σε συγκεκριμένα νούμερα, ποια είναι η διαφορά επομένω. βλέπουμε ότι έχουμε 16 εκατομμύρια γυναίκες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασία. Να, ποιο αριθμό αντιστοιχεί στο 10% τώρα, για να συνειδητοποιήσουμε τον βαθμό αυτή της ανισότητας. Ας ε, συνειδητοποιήσουμε ότι 16% είναι ο πληθυσμός μιας χώρας σαν την Ολλανδία. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το 10% διαφορά της συμμετοχής είναι σαν να έλειπε ένα κράτος μέλος που θα συνεισφέρει στην ε, οικονομία. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Είναι ένας στόχος οικονομικός και κοινωνικός. Πριν μιλήσαμε για το πώς θα ελκύσουμε την προσοχή όλων στο πρόβλημα. Σκεφτείτε, πόση είναι η οικονομική ζημία σε αυτού του χάσματος για την κοινωνία. Στη μελέτη μας προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ακριβώς το πόσο κοστίζει η ανισότητα. Πόσο χάνουμε μια που δεν μπορούμε να παράσχουμε ίδιες ευκαιρίες σε όλους για να μπουν στην αγορά απασχόλησης και οι γυναίκες. Εδώ λάβουμε υπόψη τα διαφυγόντα κέρδη, τους μη καταβληθέντες φόρους και επίσης εμ, τις ε, εισφορές που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Επομένως, θα μπορούσε να υπολογιστεί αυτή η ανισότητα ότι κοστίζει 370 δις, δηλαδή περίπου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όλα είναι η αιτησία ζημία μας, επειδή δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε, να εντάξουμε τις γυναίκες στην αγορά εργασία. Επίσης, για να συνειδητοποιήσουμε τι θα πει 370 δις. Είναι λίγο πιο κάτω από το ΑΕΠ μιας χώρας όπως το Βέλιο, χώρα στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι πληθυσμός της Ολλανδίας και ΑΕΠ του Βελγίου. Αυτό πάνε να πει ε, μισθολογική ανισότητα. Άρα είναι κολοσία η χρηματική απώλεια. Έχουμε, είπαμε, 8,2% στη Μάλτα, η Ιταλία 5,7% για την διαφορά στην απασχόληση και ε, αυτές είναι οι χώρες ε, που αντιστοιχούν σε 28 δις και μετά έχουμε την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και την Τσεχία. Επίσης το κόστος από αυτό το κενό, αυτό το χάσμα, είναι το χαμηλότερο σε Σουηδία και Λετωνία. Τώρα λάβετε υπόψη τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν αλλά δεν μπορούν. Α, τότε αν τις λάβετε υπόψη θα μειωνόταν το κόστος. Αν δούλευαν. Άρα ε, εδώ έχουμε 169 δις. Επίσης, είπαμε ότι υπάρχει και κοινωνική πτυχή στο πρόβλημα, γιατί αν κάνει δουλεύει, έχει εισόδημα και έτσι καταπολεμείται η συμμετοχή στην κοινωνία και επίσης η προσωπική ευημερία αλλά και η ευημερία της ε, κοινωνίας γενικότερα. Άρα κανείς αν συμμετέχει στην εργασία συμμετέχει σε πολλά πράγματα, πολλές δραστηριότητες και σήμερα με τα όσα λέει η μελέτη μας, ε, η απασχόληση της γυναίκας ε, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την ζωή τους. Περισσότερο αυτών που δουλεύουν παρά αυτών που δεν δουλεύουν. Υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, χειραφέτηση, γιατί έτσι υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο. Αυτό είναι επίσης πηγή ε, αυτοσεβασμού και ανεξαρτησίας. Επίσης, έτσι συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνία δεν αισθάνονται αποξενωμένε και υπάρχει μεγαλύτερο δίκτυο επαφών, γνωριμιών και συμμετέχουν και στο πολιτικό γίγνεσθε. Να, οι στόχοι μας. Και πρόσφατα έχουμε μια σειρά πολιτικών οι οποίε χαράχτηκαν τόσο ώστε να βοηθηθεί η συμμετοχή τη γυναίκα στην αγορά απασχόληση. Να, τέσσερι βασικοί τομεί, ε, όπου μπορούμε με κάποια μέτρα να κάνουμε κάτι, ε, ε, υποστήριξη τη ανθρωπής των παιδιών, πολιτική για τις ε, άδειε και περισσότερη ευελιξία στην αγορά. Πάντως, ε, να, να κάποια συμπράσματα που ε, αναφέρει με μας ότι οι πολιτικές είναι πιο αποτελεσματικές όταν υπάρχει στόχευση ακριβής ε, στο τμήμα του πληθυσμού πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η οικονομική κατάσταση οι αξίε που ασπάζεται η γυναίκα και η οικογενειακή κατάσταση. Επίση, όσον αφορά την πλαισίωση τη ανατροπή των παιδιών, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να συμμετάσχει η γυναίκα στην αγορά εργασία και είναι το, θέμα είναι το κόστο ε, τη βοήθεια για τα παιδιά, η ποιότητα και η συμβατότητα με τις, ε, το ωράριο εργασία. Επίση άλλα συμπεράσματα είναι η άδεια προς τον πατέρα προς την μητέρα. Ε, εάν είναι αμοιβόμενη αυτή η άδεια, υπάρχει ένα μικρό θετικό αποτέλεσμα. Εάν ε, αυτή η αμοιβόμενη άδεια κρατήσει πάρα πολύ, τότε μειώνεται η ένταξη της γενικής εργασίας αλλά είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ευελιξία και επίσης το πόσο ε, ο άντρας μπορεί και αυτός να δικαιούται άδειας. Επίσης ευελιξία στη δουλειά και άλλα μέτρα ε, συνδυασμού ε, δουλειά με την οικογένεια να υπάρχει κοινωνική συνένεση για όλα αυτά με το, δηλαδή ε, να συμφωνούν με αυτά οι εργοδότες να μην πρόκειται για κοινωνικό στίγμα δηλαδή να μην θεωρούν οι εργοδότες ότι η γυναίκα ζώντα τις οικογενεικές άδειες δεν είναι διαφορετική τη δουλειά. Συμπερασματικά κυρίες και κύριοι βλέπουμε ότι το χάσμα αντιστοιχεί σε 16 εκατομμύρια γυναικών που δεν έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και αυτό είναι το 10% της απασχόλησης. Δηλαδή έχουμε 370 δις ευρώ. Αυτά είναι η ζημία της κοινωνίας μας γιατί δεν μπορούμε να παράσχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η αύξηση, επομένως, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, αύξηση απασχολησιμότητας των γυναικών είναι τεράστιε μεσίε για την Ευρώπη, για το άτομο και για την οικονομία, άρα χρειάζεται ευέλικτο ωράριο εργασία, να υπάρχει ε, περισσότερη ισορροπία μεταξύ δουλειά και άλλων δραστηριοτήτων ε, και άρα θα πρέπει το ε, σχήμα, το πρόγραμμα της δουλειά, να είναι τέτοιο που να βοηθάει την ένταξη της γυναίκας. Ευκαιρίες όμως στις γυναίκες που θέλουν να δουλέψουν και άρα έτσι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασία. Πάντως μπορούμε να άρουμε αυτό το, αυτή τη διαφορά, αυτή την ε, ανισότητα, εάν όλοι ανλάβουμε έναν ρόλο τον οποίο μπορούμε να διαδραματίσουμε. Όλη η κοινωνία θα ωφεληθεί εάν γίνει πραγματοποίηση αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα Well, thank you very much. Um, is there anyone from the floor? Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο το λόγο. Σχόλια. Ναι. Υπάρχει σαφή ε, ε, διασύνδεση μεταξύ αυτού του ζητήματο και του προηγούμενου. Ε, τα τελευταία αυτά σημεία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την φροντίδα του παιδιού χρειάζονται τα στοιχεία που να αποδεικνύουν σαφώς ε, ότι χρειάζεται αυτή η σωστή φροντίδα για τα παιδιά, αυτή η υποστήριξη έχει πολύ μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο αυτό που να επενδύσουμε σε μια κατασκευή και σε μια υποδομή. Γιατί όταν μιλάμε για υποδομή, μιλάμε για γέφυρες, Και βεβαίως ε, οι κοινωνικέ υποδομέ είναι η φροντίδα των παιδιών αλλά και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν είχα βεβαίω την ευκαιρία να εξετάσω την έκθεση αλλά πραγματικά θα εκτιμούσα ιδιαίτερα να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τα απτά ε, τα οποία να μας βοηθούν στην πολιτική μας στόχευση. Ακόμα μερικά σημεία για το θέμα του χάσματος των αμοιβών στον, στο τομέα της απασχόλησης. Βεβαίως ε, χρειάζονται παρεμβάσεις από το σχολείο και μετά για να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες στους συγκεκριμένους αυτούς κλάδους ε, θα έχουν παρουσία, θα έχουν πρόσβαση. Αυτό ισχύει και για την αγορά εργασίας, διότι υπάρχει πρόβλημα και στα 20 και στα 30 σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς. Ε, και βεβαίως ε, αυτό αφορά και το κενό στις αμοιβές Και το τελευταίο, αναφερθήκατε στην τελευταία διαφάνεια, στην πρώτη τελευταία βασίλισσα διαφάνεια, ε, να υπογραμμίσουμε εκ νέου ότι το θέμα της οικογενειακής φροντίδας δεν είναι ευθύνη μόνο της γυναίκας. Ε, πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία του ρόλου του πατέρα ή του οποιοδήποτε περιπτώσει άλλου μέλους της οικογένειας για να έχουμε έτσι και την ευρύτερη εικόνα. Δεν μπορούν οι γυναίκες να κάνουν τα πάντα συνεχώς. Προσπαθούμε. Ορισμένε φορές ε, ε, πετυχαίνουμε πολλά, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι η υποστήριξη ε, στους τομείς αυτούς πρέπει να έρθει από πολλά πρόσωπα. Μάλιστα. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Ναι, εν συντομία θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τα ερωτήματα. Ναι, ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, γίνεται αυτό το εγχείρημα να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε το κόστος ε, του χάσματος ε, να δείξουμε ότι δεν αρκεί να επενδύσουμε σε γέφυρες, πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους, να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους για να έχουμε πραγματικά μετρήσιμα εργαλεία. Ε, το να χτίσουμε ένα, μια γέφυρα δεν το κάνει αυτό. Και βεβαίως, ε, προφανώς η ευθύνη είναι κοινή. Πρέπει να είναι μοιρασμένη ανάμεσα στο ανδρικό και στο γυναικείο φύλλο. Έκανα και μια άλλη μελέτη για τις ανάγκες των ε, των νέων που δεν ούτε, εργάζονται ούτε φοιτούν και πολλές, το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο μέρος των, των αναγκών έχουν να κάνουν με τις ευθύνες ε, των, των, οικογενειακές. 92% είναι γυναίκες. 2,7 εκατομμύρια γυναίκες, 300.000 άντρες. Ε, πρέπει να ξεκινάμε λοιπόν από το σχολείο και από εκεί να το πιάσουμε διότι σε πολύ μικρές ηλικίες ξεκινάει το πρόβλημα των ίσων ευκαιριών. Αναφερθήκατε και στην φροντίδα προς τους ηλικιωμένους. Είναι και ένας άλλος τομέας. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, διότι υπάρχει μια τάση ε, στο επίπεδο απασχολησιμότητας ε, που σχετίζονται άμεσα με τη φροντίδα και των ενηλίκων και των παιδιών. Ναι, το άλλο που είπα έχει να κάνει με την τεχνολογία, ε, τη μηχανική, τα μαθηματικά, τις επιστήμες γενικότερα και ότι πρέπει η εκπαίδευση των κοριτσιών ε, να είναι τέτοια που να τους δίνει το δικαίωμα, πάνω να έχουν την πεποίθηση ότι έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στην καριέρα τους και σε αυτές τις επιστήμες. Αυτό ήταν το δεύτερο που ανέφερα. Πολύ ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι από αυτού? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει, υπάρχουν διακρίσεις. Ε, αυτό οδηγεί και σε διακρίσεις ε, και στην εκπαίδευση και στην αγορά Πρέπει να το ανοίξουμε αυτό το θέμα, να πάψουν οι διακρίσεις να γίνουν αυτές οι, οι σπουδές πιο ελκυστικές και να δώσουμε και την ευκαιρία συμμετοχής. Ιδάλλως δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο της διάκρισης που στη συνέχεια βεβαίω τη βρίσκουν μπροστά του οι γυναίκε και στην αγορά εργασία. Μάλιστα, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μασκερίνη όλους ιδιαίτερω για την πραγματικά ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση. Ελπίζω όλα τα μέλη να τη λάβουν υπόψη του. Περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχείο. Ένα τελευταίο θέμα πριν πάμε στα διάφορα που είναι η Σύνος Κορυφής των Γυναικών στην Πολωνία. Ε, δεν ξέρω αν η Κλέρα έχει να, να πει κάτι από αυτού. Ε, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, ε, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε το σχετικό κείμενο της έκθεσης δηλαδή εγκρίνεται λοιπόν και φτάνουμε τώρα στα διάφορα δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα πολύ ωραία ολοκληρώνεται λοιπόν η συνάντησή μας σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας